Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ όσοι φεύγουν με ησυχία. Γιατί τώρα ξεκινάμε τις ε, επεξηγήσεις ψήφου. Πριν από αυτό, να σας πω πως ε, ξεκινάμε με τις επεξηγήσεις ψήφου που δεν ακούστηκαν χθες και μετά θα περάσουμε στις σημερινές επεξηγήσεις ψήφου και έχω λάβει και αιτήματα για προφορικές επεξηγήσεις ψήφου. Η συνεδρίασή μας δεν μπορεί να πάει πέρα από τις δύο η ώρα. Έχουμε λοιπόν μία ώρα. Και οι υπόλοιπες γραπτός. έχει κυρία Νίνα Γκίλ για ένα λεπτό. Ο κύριος Πόλτσακ, ούτε ο κύριος Πόλτσακ είναι εδώ. Η κυρία Μορβάη λοιπόν. Για ένα λεπτό. Με μικρόφωνο, με μικρόφωνο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόλτσακ, για ένα λεπτό. Ναι, ναι, έχετε το λόγο. Ε, δεν ήταν στην αίθουσα ο κύριος Πόλτσακ, ε, σας έδωσα το λόγο, αλλά εντωμεταξύ ήρθε και τώρα θα λάβει εκείνος το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαρά υπερψήφισα την έκθεση για την πολιτική συνοχής. Γιατί ψήμου αντιδρά πάρα πολύ καλά στην κατάσταση. Γιατί αντιδρά πάρα πολύ καλά στην κατάσταση των πιο ασθενών περιοχών και όσων χρειάζονται την στήριξή μας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Επίσης πρέπει να εστιαστούμε στο να στηρίξουμε τις βασικές μας περιοχές, ε, εκεί όπου βρίσκεται ο πληθυσμός, αλλά και άλλες περιοχές που έχουν κάποια ανάγκη. Για το μέλλον λοιπόν θα πρέπει να εστιαστούμε στην αηφόρο ανάπτυξη, γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το σημαντικότερο κομμάτι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, έκθεση για τη συνοχή, συνοχή προφανώς την υπερψήφισα, γιατί εγώ κατάγομαι από μια χώρα που είχε μείνει πίσω και βεβαίω ε, το ζήτημα είναι πώς θα δυναμηθούν αυτά τα λεφτά, γιατί αυτή τη στιγμή η Ουγγαρία δεν ε, θεωρεί ότι θα μπορέσουμε έτσι να αντισταθμίσουμε τις διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το ένα είναι... Οι φόβοι μας, τους οποίους είχαμε ήδη πριν από την ε, ένταξη. Και από την άλλη ότι μας χτυπάνε από δύο μεριές. Έχουμε τις παγκοσμιοποιημένες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις και από την άλλη οι δικοί μας ολιγάρχες. που μοιράζονται τον πλούτο της ε, Ουγγαρίας και εκμεταλλεύονται τις δυνάμεις ε, της χώρας μας. Ε, αυτή είναι η κατάστασή μας. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Έχετε το λόγο κυρία Μακοβέη. microfon. Da, da, da, am spus că primele vor fi cele care sunt de ieri. Ε, η, δύο, η πρώτη ήταν από τις χθεσινές επεξηγήσεις ψήφου. Δεν θέλει η κυρία Μακοβέη το λόγο. Πολύ ωραία. Ο κύριος Έθωριτς απουσιάζει. Ο κύριος Μπόγκοβιτς και και εκείνο απόν. Η κυρία Μάλετιτ. Απούσα. Ο κύριος Κέλλη. Και εκείνος απουσιάζει. Κύριε Μαμίκινς, είστε εδώ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά υπερψήφισα την έκθεση Deutsch γιατί και από λατωνικής πλευράς και εμπειρίες διαπιστώνουμε ότι δύο διαδικασίες εκτιλήσονται παράλληλα. Η ανάπτυξη των ε, πιο μειονεκτουσών περιοχών και η εμπορική πολιτική, ε, πολιτική ανταγωνισμού. Βέβαια το σύστημα μέχρι στιγμής ε, ήταν ανεπαρκές και ατελέσφορο. Πρέπει να μειώσουμε το αναπτυξιακό κενό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη έκθεση θα συμβάλλει στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάρκιν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Προέδρε. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η έκθεση. Προωθεί την επένδυση για απασχόληση και ανάπτυξη τη περιοχή τη Ευρωπαϊκή Ενώση. πολύ συχνά βλέπουμε ότι επενδύσει επικεντρώνονται στι πόλει ε, και στι αστικέ περιοχέ, χωρί να λαμβάνουν υπόψη την ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχυρέ χώρε χρειάζονται ισχυρέ περιφέρειε και η ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ισχυρέ περιφέρειε. Η πολιτική συνοχή στο βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να προωθήσουμε τι ισχυρέ περιφέρειε και δίνουμε τώρα τίτλο υπολογισμού. Αν θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη απασχόληση στην Ήπεθρο και στι περιφέρειε, τότε θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε πρόσβαση σε περιφερειακή ευρυζωνική και ευρυζωνική στην Ήπεθρο. Μπορεί να έχουμε ψηφιακή ένωση αν δεν έχουμε πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία σε όλη την ένωση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην Ιρλανδία, Φερρυπίν. Δεν έχουμε πρόσβαση στη ψηφιακή τεχνολογία σε όλη τη χώρα. Συνεπώ, η ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη και η ισότητα δυνατοτήτων, αυτέ οι εκφράσει δεν έχουν νόημα μέχρι ότου να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Νίνα Γκίλ έχει το λόγο, δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Πόσπισιλ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή όσον αφορά την αξιολόγηση του έτους για την ενεργογύρανση Είμαι πεπισμένος ότι οι ηλικιωμένοι είναι σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού μα και θα αυξηθεί το ποσοστό στο μέλλον. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την ενεργό αυτή γύρανση, να στηρίξουμε τι δεξιότητε που έχουν οι ηλικιωμένοι μα πολίτε και να βελτιώσουμε και τι γνώσει που έχουν σαν αφορά του υπολογιστέ. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι οικογένειε για να μπορούν να εντάξουν στη ζωή του του ηλικιωμένου μπορείτε να βρείτε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη μέρημνα για τους ηλικιωμένους. Αυτές οι διαφορές δεν αφορούν μόνο τι συντάξει και τα κοινωνικά επιδόματα, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν οι ηλικιωμένοι για να μπορούν να ζουν. Ελπίζω λοιπόν αυτό το πρόγραμμα για την ενεργογύρανση ε, θα προωθηθεί και δεν θα λησμονήσουμε τα πάντα μετά την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Αυτή τη στιγμή ακούμε τις επεξηγείς ψήφου επί της εκθέσεως Κούκαν, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο κύριος Μπόγκοβιτς έχει το λόγο. Όχι, όχι, είναι η σειρά του κυρίου Μπόγκοβιτς, αλλά απουσιάζει. Οπότε κυρία Ζάμπορσκα, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αλληλεγγύη προς τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η έκθεση Κούκαν έθιξε το ζήτημα το ύψος των συντάξεων των γυναικών. Εδώ πέρα απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα. Είναι άδικο και λάθος να τιμωρεί η κοινωνία μας τις γυναίκες, χωρίς οποίες δεν θα υπήρχε η νέα γενιά. Οι γυναίκες αναθρέφουν τις νέες γενιές για ευθύνη και αλληλεγγύη και βεβαίως ταυτόχρονα εκτιμώ πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να λάβει υπόψη τη χρονιά της ελεγγύης και της ενεργογύρανσης. Κύριος Κέλλη, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Με χαρά στήριξα την έκθεση Κούκαν, λέει ο κύριος Μαμίκινς, γιατί γεγονό είναι πως ο πληθυσμός γυράσκει και χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Το 2015 η μέση ηλικία της Ευρώπης ήταν πάνω από το 2050. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν στην οικονομία, την κοινωνική σφαίρα και την εκπαίδευση. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα βιβλία που εξηγούν ε, το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες ε, απασχόλησης αλλά όλα αυτά ειδικά στη χώρα μου ε, την Λετωνία δεν γίνονται και άρα απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό Και εγώ ψήφισα υπέρ τη έκθεση για την ενεργό και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Όταν λέμε ενεργογύραση ε, εννοούμε σωστή υγεία, μη διακριτική μεταχείριση, πρόσβαση σε, στην παιδεία των ανηλίκων, μεταφορές, ε, υγεία και φυσικά θέματα συνταξιδοτικά. Η έκθεση όμως αυτή δεν μιλά μόνο για την ενεργογύρανση αλλά και για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στεναρό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει το κατά πόσο είναι εφικτό και τι προστιθέμενη αξία επιφέρει ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί ελάχιστο εισόδημα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που διαβίουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Βέβαια το θέμα αυτό, το ελάχιστο εισοδήματος, είναι εθνική αρμοδιότητα. Αν όμω ένα ευρωπαϊκό εργαλείο έχει κάποια προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να το μάθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, αναφέρουμε το πόσο μας λυπεί η κατάσταση όταν η απασχόληση γίνεται όλο και πιο επισφαλής και αυτό επηρεάζει όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως τους νέους. Ο κύριος Πόρτσακ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ υπερψήφισα την έκθεση Κούκαν γιατί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και από τις πιο σημαντικές ε, αρχές μας ε, προκειμένου να συμβάλλουμε και να στηρίξουμε την ε, υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Η γύρανση είναι γεγονός γιατί οι δημογραφικές εξελίξεις το βεβαιώνουν. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τους νέους αλλά και τους ε, ηλικιωμένους ώστε οι οικογένειες μένουν ενωμένε όσο περισσότερο γίνεται. Έχουμε πολλές υπηρεσίες που βοηθούν τις οικογένειες ε, να κρατήσουν τους ηλικιωμένους τους και να μην τους βάζουν στα γυροκομεία. Νομίζω αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα βέρτιση των πρακτικών και αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Πάμε στην έκθεση κάμπ. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόπεθ. Δεν είναι στην αίθουσα. Η κυρία Σίμερτζιλ δεν είναι παρούσα. Ο κύριος Κέλλη απουσιάζει. Κύριος Μάμικινς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα αυτή την έκθεση. Θεωρώ ότι η άποψη που εκφράζει είναι σημαντικότατη για την 21ο αιώνα. Ο στόχος της Λευκή Βιβλού για τις μεταφορές είναι να, να έχουμε ένα στρατηγικό όραμα, να έχουμε αποτελεσματικά μεταφορικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και εφόσον πρέπει να επανεκκινήσει η οικονομία μας, πρέπει να βασιστούμε στο μεγάλο τεράστιο ρόλο που μπορεί να παίξουν οι μεταφορές. Ζητήσαμε να λάβει συγκεκριμένα βήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους, ώστε το στατηγικό όραμα που προανέφερα να μπορεί να υλοποιηθεί με αυτό τρόπο και να έχουμε πραγματικά διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και θα είναι χρησιμότατο κάτι τέτοιο για μας στο μέλλον. Λούνγκρεν, ο κύριος Λούνγκρεν απουσιάζει. Επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Βόζενμπεργκ. Η κυρία Ζόιντροβα έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την έκθεση Βόζενμπεργκ διότι πιστεύω ότι η συγγήτρια έκανε πολύ καλή δουλειά και συμφωνώ με το περιεχόμενο. Μιλάμε για την ισότητα των φύλων, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι αυτή η ισότητα δεν αποτελεί συχνά πραγματικότητα. Υπάρχουν στερεότυπα. Δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες σε διάφορους τομείς όπως είναι τεχνολογία και οι επιστήμες. Στόχος της εκθέσεως είναι να αρθούν η αόρατη φραγμή για τις γυναίκες που τις εμποδίζουν να κάνουν καριέρα. Θα θέλαμε εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κυρίως στον τομέα των επιστημών. Υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν δυνατότητα στις γυναίκες να επιστρέψουν στην επαγγελματική του ζωή χωρίς να χάσουν την επαφή με τον τομέα της μελέτης τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζιτνάνσκα απουσιάζει. Η κυρία Φορέντσα. Ε, Εγώ υποστήριξα το κείμενο αυτό που μας καλεί να δούμε πόσο υπάρχει αυτός ο αόρατος στόλος που εμποδίζει τις γυναίκες να κάνουν πανεπιστημιακές καριέρες ή σε τον ερευνητικό τομέα. Αόρατα φράγματα. Προσωπική εμπειρία είναι αυτή. Ξέρω μία ε, είμαι μια ερευνήτρια ερευνητη ορισμενου χρόνου και υπό αυτή την ιδιότητα μιλώ. Έχει καθήκον η Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει τέτοια εμπόδια, εμπόδια που οφείλονται σε διακρίσεις ε, με βάση το φύλλο, έμφυλες διακρίσεις ε, που υπάρχουν στον πανεπιστημιακό τομέα θα πρέπει να πούμε σαφέστατα ότι η διαδικασία προσωρινής εργασίας στο Πανεπιστήμιο έπληξε πάνω από όλα τις νέες γυναίκες και τις νέες ερευνήτες αυτή η αβεβαιότητα. Πρέπει να αλλάξει ριζικά η κατάσταση, θα πρέπει να δράσει ριζικά η Ένωση για να μην υπάρχουν αυτού του διακρίσεις και θα πρέπει να επανέλθει η χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια που είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο για να αντιμετωπιστούν οι ε, έμφυλες διαφορές. Σα σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ήμουν ερευνητή κάποτε. Κυρία Νίνα Γκίλ έχει τώρα το λόγο, δεν είναι στην αίθουσα. Πάρκερ, δεν είναι εδώ. Η κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τις γυναίκες στα πανεπιστήμια θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στην κατάσταση στην Ιρλανδία όπου το δικαστήριο για θέματα ισότητας αποφάσισε ότι για την περίπτωση της Μισελ Σκέφινγκτον υπήρχε άμεση και έμεση διάκριση κατά των γυναικών για να προαχθεί σε επίκουρο καθηγητή. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Μάλιστα το 2009 μόλις 10% των ανώτερων ε, θέσεων καθηγητών πανεπιστημίων και μάλιστα μετά τη Μάλτα η κατάσταση είναι χειρότερη στην Ιρλανδία. Ναι, υπήρξε μία αντίδραση, αλλά παραμένει άνηση. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες των δύο φύλων, να υπάρξει προϋπολογισμός για το θέμα αυτό, αυξημένη συμμετοχή των γυναικών και σχέδια ισότητας ως προϋπόθεση χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ η κυρία Μορβάη. Υποστήριξα την έκθεση για τις καριέρες ε, των γυναικών. Γιατί το έκανα αυτό. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Συγκλονιστικό. Αυτή τη στιγμή πάνω από τις μισές ε, από είναι γυναίκες. Όταν μιλάμε όμως για Πριτάνης, ε, μόνο 10% είναι γυναίκες. Το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων και των γυναικών με διδακτορικά. Δυστυχώς πάρα πολλές από αυτές παρατάνε την επιστημονική τους καριέρα αφού λάβουν το διδακτορικό τους, συνήθως λόγω παιδιών. Δεν είναι φυσικό. Και δεν είναι φυσικό να υπάρχουν τόσες λίγες ε, Περιτάνεις. Πρέπει να ερευνήσουμε το ζήτημα και σας καλώ να μου στείλετε επιστολές και email. Μάλιστα. Μπίχνερ. Βεβαίως η ίση μεταχείριση και αξιολόγηση των δύο φύλων είναι βασικό θέμα στο οποίο κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση. Αλλά στις δύο εκθέσεις, ε, Ροντρίγκε και Βόζενμπεργκ, οπωσδήποτε δεν θα καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Γιατί οι σπουδές στις ε, φυσικές επιστήμες δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίζει κανείς λόγω διαφήμισης. Οι σπουδές είναι σκληρή δουλειά. Δεν είναι περίπατος και ε, είναι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάλογη κλίση. Βλέπουμε τον ψηλό αριθμό ατόμων ε, που τα παρατάνε. Γιατί για να περατώσει κανείς τις σπουδές του πρέπει να στρώσει κόλλο, κάτι το οποίο οπωσδήποτε δεν θα κάνουν όσοι πίστηκαν από μια διαφήμιση. Και βεβαίως το να διακόψει κανείς σπουδέ του σημαίνει ότι χάνει χρόνο από τη ζωή του και πολλά χρήματα. Γι' αυτό θεωρώ πως οι εκθέσεις αυτές είναι ανεύθυνες και δεν βοηθούν τις νέες γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάχθηκα υπέρ τη ε, της έκθεσης γιατί είναι κρίμα που μετά από τόσες συζητήσεις και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0. Επιπλέον οι γυναίκες καθημερινά ξεπερνάνε τα όρια τους, καταρρύπτουν ρεκόρ, δημιουργούν νέες ε, ευκαιρίες αλλά πάντα υπάρχει η εντύπωση ότι αξίζουν λιγότερο από, ε, από τους άνδρες. Βρίσκουν κλειστές τις πόρτες και της εργασίας και των προαγωγών ε, ενώ συχνά είναι πιο μορφωμένε από του άντρε που πολύ εύκολα περνάνε από τι πόρτε αυτέ. Η γυάλινη οροφή στηρίζεται στι προκαταλήψει που δημιουργήθηκαν από την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να ενθαρρύνουμε τι γυναίκε, να τι εμψυχώσουμε, να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί είναι ικανέ να επιτύχουν πολλά, να συνδυάσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή και να φτάσουν σε ηγετικέ θέσει. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίσους όρους για τους άνδρες και τις γυναίκες στην εργασία, στους μισθούς και στις προαγωγές. Ε, βέβαια η λύση δεν βρίσκεται στις ποσοστώσεις, αλλά στην αλλαγή της νοοτροπίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου της έκθεσης για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, μήπως κάνω λάθος. Α, όχι, προηγείται η έκθεση Ροντρίγκε. για τη χειραφέτηση των γυναικών μέσω της παιδείας. Η κυρία Φων Στόρχ απουσιάζει, η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η έκθεση για τη χειραφέτηση των ε, γυναικών ε, δυστυχώς δεν με βρίσκει σύμφωνη. Παρόλο που ο τίτλος είναι καλός, η έκθεση βρήθη προβλημάτων και σημείων που αντιστρατεύονται βασικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταστρατηγούν ε, το δικαίωμα στη πρόσβαση στην παιδεία, στην σεξουαλική υγεία Ουσιαστικά η έκθεση δεν προσφέρει τίποτα καινούριο, ούτε κάποιες ε, ε, απτές και χειροπιαστές προτάσεις. Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι, αλλά οι ευκαιρίες είναι διαφορετικές. Σίγουρα η υγιής παιδεία είναι η βάση μιας υγιούς κοινωνίας και πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη, αλλά δεν είναι σωστός ο τρόπος που προτείνει η έκθεση. Για παράδειγμα, προτείνεται υποχρεωτική εισαγωγή της ε, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, κάτι που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Χαίρομαι πάντως που δεν είναι δεσμευτικό αυτό το κείμενο και δεν, μπορούν, δεν χρειάζεται αυτόματα να το δεχτούν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τζιμπνάσκα, απουσιάζει. Η κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ με μεγάλη ικανοποίηση ενέκνα την έκθεση. Τη στήριξε ένθερμα. Διότι εδώ στο κοινοβούλιο, στην αίθουσα αυτή, είδαμε ότι υπήρχε κάποια σύγχυση όσον αφορά τη θεωρία του φίλου, των φίλων και την εκπαίδευση με βάση αυτή. Εγώ νομίζω ότι αυτό ο τρόμος που επικράτησε συζητήσει ήταν άλμα στο μεσαίωνα. Η έκθεση που εγκρίθηκε ε, επιτρέπει να αποφύγουμε το άλμα προς το πίσω. Λοιπόν, η, η, η σεξουαλική αυτή αγωγή στα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική της Ένωσης κατά της ε, διάκρισης με βάση το φύλλο, κατά του σεξισμού, κατά της ομοφοβίας. Λοιπόν, με μεγάλη ικανοποίηση ε, χαιρετίζω την έγκριση της εκθέσεως. Λοιπόν, και τα, οι μελέτες των θεμάτων των φίλων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα που διδάσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Νίνα Γκίλ δεν είναι εδώ. Η κυρία Πάρκερ δεν είναι εδώ. Η κυρία Μορβάη το ίδιο. Η κυρία Ζαμπόσκα. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. práve Σας ευχαριστώ. Βεβαίω θα πρέπει να μπορεί η κάθε οικογένεια να επιλέγει την εκπαίδευση των παιδιών της για να μην υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Οι γονείς είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών και αυτό είναι το δικαίωμα και στην διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου τέτοιοι όροι όπως ε, φύλο, gender, δεν υπάρχει ορισμός για αυτά τα πράγματα και πρέπει να οριστούν. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες κάθε φορά. Δεν είναι σωστός αυτός ο όρος για το πλαίσιο στο οποίο το χρησιμοποιούμε. Η ταυτότητα του φίλου για την οποία μιλάει αυτό το ψήφισμα δεν έχουν βάση στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα και δεν έχουν ε, θέση στην υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών. Είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κατά των ηθών μας. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση για την παιδεία σε αυτό το τομέα πρέπει να μας ξυπνήσει το Κοινοβούλιο. Δεν θα μπορούμε να λησμονήσουμε τη Μαλάδα και Σαφάη και την ομιλία που έκανε για το πόσο μέσω της παιδείας αποκτούν ισχύ τα κορίτσια. Η γνώση είναι ισχύς και ζούμε σε οικονομία της γνώσης. Υποστηρίζω την πρόταση της εκθέσεως να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τα κράτη-μέλη να την επικυρώσουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για την ισότητα των φύλων όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα χαράς υποστηρίζω ε, την εκπαίδευση όσον αφορά το φύλλο και την εκπαίδευση όσον αφορά τις σχέσεις και ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη μελη να κάνουν, να προβούν σε υποχρεωτική ε, εκπαίδευση στον τομέα, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει όμως να είναι ανάλογη εκπαίδευση με την ηλικία. Οι περισσότεροι να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό με όλα τα θετικά και αρνητικά που συνεπάγεται αυτό. Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα τα παιδιά με τη σωστή εκπαίδευση για την ηλικία τους και για τις σχέσεις εκπαίδευση. Διαφορετικά δεν έχουν σωστή ε, ισχύ και δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτά που βλέπουν και αυτά που ακούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούχνερ. Έφυγε. Κύριε Πετήρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η έγκριση της έκθεσης αυτής αποτελεί την της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Γι' αυτό και την καταψήφισα. Τέτοιες ιδεολογίες ανήκουν στο παρελθόν ε, αλλά οι σοσιαλιστέ φαίνεται ότι επιχειρούν να μα τι επιβάλλουν εκ νέου. Το χειρότερο είναι ότι το κάνουν υπό το πρόσχημα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Με την έκθεση αυτή στερούμε από του γονείς τη δυνατότητα να αποφασίσουν για την ανατροφή των παιδιών τους και από τα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν τα σχολικά του προγράμματα. Ε, διαρωτόμαστε λοιπόν τι πρόκειται να ακολουθήσει και πρέπει να το διαρωτηθούμε αυτό, γιατί φαίνεται ότι μερικοί ευρωβουλευτές δεν γνωρίζουν ε, τις θέσεις και τις αξίες των ε, ψηφοφόρων τους. Εγώ ψήφισα κατά γιατί η έκθεση αυτή αντιβαίνει στην Ευρώπη στην οποία πιστεύω. Γιατί είμαι υπέρ μιας Ευρώπης στην οποία έχουν θέση και ανθρώπινες αξίες, κάτι που αντιστρατεύεται η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ στις επεξηγήσεις ψήφου των σημερινών ψηφοφοριών. Πρώτα, επεξηγήσεις ψήφου για το ψήφισμα μετανάστευσης και προσφύγων στην Ευρώπη. Ο κύριος Πόσπισιλ, γιατί η κυρία Φορέντζα απουσιάζει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση, γιατί κατά τη γνώμη μου ε, δράζεται σε εσφαλμένη φιλοσοφία που προβλέπει ότι η Ευρώπη μπορεί να λύσει το μεταναστευτικό κατανέμοντας τους μετανάστες με βάση τις ποσοστώσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που υπολογίζονται με αδιαφανή κριτήρια. Πιστεύω ότι οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής της χώρας προορισμού, ε, προορισμού τους ε, και εκεί να πηγαίνουν και τότε η χώρα υποδοχής να, να αποφασίζει με βάση το διεθνές δίκαιο αν θα τους δεχτεί ή όχι. Είμαι υπέρ τη στήριξης, οικονομικής υποστήριξης των προσφύγων ή ε, των μεταναστών, αλλά διοικητικέ λύσει ε, του τύπου υποχρεωτικό ποσοστό δεν πρόκειται να διορθώσουν τίποτα. Και στην Τσεχία όλο και περισσότερο ακούγονται φωνές κατά του Σέγγεν. Ε, όσο περισσότερο θα αυξάνεται η λαθρεία μετανάστευση στην Ευρώπη, τόσο θα πολλαπλασιάζονται οι πολέμοι του Σέγγεν. Θέλουμε διαφορετική πολιτική από αυτή που θετήσαμε σήμερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Αποφάσισα να υπερψηφίσω την έκθεση, λέει ο κύριος Κρέσπο, γιατί σε τελική ανάλυση ε, συμπεριέλαβε μία τροπολογία που υποβάλαμε με το παράδειγμα των πόλεων ε, καταφύγια που ελπίζουμε να γίνουν υπόδειγμα στην Ευρώπη. Η Ισπανία της ε, προέβλεψε το μοντέλο αυτό και τελικά όταν οι κυβερνήσει αμέλησαν να αναλάβουν μέτρα, οι, ε, οι πολίτες, ο κόσμος ε, δημιούργησε τη, την ε, ροπή για να δημιουργηθούν ε, πραγματικά μέτρα ανθρωπιστικά. Χθε μας είπε μεγάλα λόγια ο κύριο Γιούγκερ για την Ευρώπη, για την αλληλεγγύη. Ωραία όλα αυτά τα λόγια, αλλά είναι ε, λόγια απλώ του αέρα. Πρέπει να συνοδευτούν από πράξεις, γιατί οι μόνες πράξεις που βλέπουμε είναι οι, φρα... φράχτες και που υψώνονται όλο και πιο ψηλά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πολιτικές από τη βάση για να στηρίξουμε ε, την αλληλεγγύη και να οικοδομήσουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζντάνοκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Ε, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο μα χωρίς ρίζες. Το πρώτο πρώτο εκτιμώντας λέει πως ε, ένας ε, πρωτόγνωρος αριθμός ανθρώπων ζητούν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω συγκρόσεων κτλ. κτλ. Μα αυτή η αστάθεια είναι συνέπεια τίνος πράγματος. Πού είναι η αιτία. Το ψήφισμα δεν δίνει την απάντηση αυτή. Πολλοί από αυτούς ε, τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπουργοί ε, δημιούργησαν ε, την αστάθεια αυτή σε Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκ και τώρα είναι σε αυτή την αίθουσα. Τώρα θένε να μεταθέσουν την προσωπική ευθύνη στους ώμους όλων των φορολογουμένων. Οπωσδήποτε να είμαστε ανθρώπινοι απέναντι στους πρόσφυγες, αλλά η ανεύθυνοι αυτή η πολιτική δεν αξίζουν ανθρώπινη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ στήριξα το ψήφισμα αυτό Πρόκειται για μια κατεπίγουσα αντίδραση σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν μπορούμε να γυρνάμε την ε, πλάτη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φτάσει σε μια συνεκτική θέση. Θεωρίζαν πως η οικονομική κρίση ήταν δυσκολία. Και ήταν. Αλλά αυτή η κρίση είναι ακόμη μεγαλύτερη ε, δοκιμασία. Είναι ζήτημα ανθρωπισμού. Εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο Πολ Φράνσις κάθε ενορία να πάρει από έναν πρόσφυγα και βεβαίως ε, χαιρετίζω και τους ΜΚΟ που καλώς ορίζουν ε, πρόσφυγες. Αλλά πρέπει να υπάρξουν και νόμιμες οδημία μπλε κάρτα, αλλά και να επιστρέψουμε πίσω τους οικονομικούς μετανάστες που έρχονται παρανόμως πρέπει να συνεργαστούμε με την Αρμοστία του για τους πρόσφυγες για να φτιάξουμε ε, στρατόπεδα φιλοξενίας, χώρους φιλοξενίας στη Βόρεια Αφρική και επίσης ασφαλείς ζώνες. Μπάλτσο. Σας ευχαριστώ. Το ψήφισμα όσον αφορά τη μετανάστευση αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα και την κρίση της μετανάστευσης. Βλέποντας το ψήφισμα και τις δηλώσεις κάποιων επικεφαλής ηγετών κρατών, βλέπουμε ότι είναι μια πρόσκληση ανοιχτή προς τους πρόσφυγες. Είναι παράνομοι μετανάστες αυτοί, όχι ε, πρόσφυγες. Πάνω από 195.000 ε, τα σύνορα στην Ουγγαρία, με παράνομο τρόπο και αυτό δημιουργεί αναταραχή στον τόπιο πληθυσμό. Η Ουγγρική κυβέρνηση ε, διε, συμμορφώνεται με απερχιωμένους κανονισμούς που θα πρέπει να απορριφθούν. Μόνο έτσι μπορεί να διαφυλάξει την κυριαρχία της Ουγγαρίας και των συνόρων Σέγγεν Ουγγαρία. Θα πρέπει βέβαια να ληφθούν υπόψη ανθρωπιστικές πτυχές στην επίλυση της κρίσης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη βασική αρχή ότι η Ευρώπη ανήκει στους Ευρωπαίους. Η κυρία Μίτσι έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που συνέβησαν στη Λαπεδούσα, ε, παρόλα αυτά και παρά τα ναυάγια και τις χιλιάδες ζωές που χάθηκαν, μένουμε μόνο στα λόγια. Χθε το είπε ο κύριος Γιούγκερ και το χειροκρότησα. Γιατί πολλά λόγια λέμε, γεμίζουμε το στόμα μας με ωραίες λέξεις και ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή ε, γυναίκες και παιδιά δίνουν μάχη για τη ζωή τους, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τις διώξεις. Ε, η Ευρώπη φαίνεται ότι είναι ένας χάρτινος τίγρης ε, και ε, δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων και στην υποχρέωση που έχει να δείξει αλληλεγγύη. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς την αξιοπρέπειά τους γιατί την αξίζουν και φυσικά να λάβουμε υπόψη το μέγεθος των χωρών που θα υποδεχθούν τους μετανάστες. Ευχαριστώ κύριε Μαμίκης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν πλήρη μεχανισμό για να μπορεί να αντιμετωπίζει ε, το πρόβλημα των προσφύγων. Διότι αυτό είναι ένα θέμα που θα παραμείνει μπροστά μας. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη προσέγγιση, όχι γενική. Θέλουμε κοινή μεταναστευτική πολιτική και συγκεκριμένη πολιτική για τους πρόσφυγες. Η κρίση λοιπόν μπορεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν δεν κινηθούμε μαζί θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα να επιληθεί. Έχουμε την οικονομική κρίση και τώρα παρουσιάστηκε και η κρίση αυτή με τους πρόσφυγες. Κινούμεθα αργά προς μια κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου και πρέπει αυτό να ελοποιηθεί, διαφορετικά θα αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα. Κύριος Χάναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση για τι ποσοστώσει για τι πρόσφυγε, αλλά δεν είναι βιώσιμη ούτε πλευρά ηθική ούτε πρακτική. Ποια είναι η ηθική αντίρρηση. Ήδη ο κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε του πρόσφυγε τη Συρία, αντί να στηρίξουμε το Σέγγεν, θα του παίρναμε από τα στρατόπεδα κατευθείαν. Όταν ήδη κάναν στι σχετικά ασφαλεί χώρε Ευρωπαϊκή Ενώσεω και κάνουν το ταξίδι, τελικά βραβεύουμε του διακινητέ. Και υπάρχει και πρακτική αντίρρηση. Δεν μπορεί να έχει ποσοστώσει και την αρχή τη ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Κάποτε αυτοί οι πρόσφυγε θα αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα και τα δύο είναι ασύμβατα μακροπρόθεσμα σαν αρχέ. Το Σέγγεν όπω το ευρώ ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούσε να επιβιώσει. Δεν ήταν ανθεκτικά. Λειτουργούσαν όταν ήταν καλό ο καιρό και είχαν, υπήρχε λιακάδα, όταν οι καταιγίδε κατέρευσαν. Τεράστιε φιλοδοξίε η Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν συντρίμια και μένουν τελικά σαν μνημεία στην έρημο, σαν ερήπια στην έρημο όλες αυτές τις φιλοδοξίες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μόρβαη απουσιάζει. Η κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Και πάλι δεν μπόρεσα να ψηφίσω υπέρ, γιατί και πάλι ε, βρήκα συστάσεις ή εκκλήσεις ε, για υποχρεωτικές ποσοστώσεις ό,τι αφορά την κατανομή των προσφύγων. Αυτό είναι ένα μοντέλο που μας λένε ότι θα πρέπει να γίνει η βασική στερεότυπη λύση. Κατά τη γνώμη μου κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει πάντα να έχουν την δυνατότητα να καταλήγουν σε συμφωνίες ε, μεταξύ τους. Δεν μπορεί κάποιος να τους υπαγορεύει πόσους ε, πρόσφυγες θα υποδεχτούν. Ακόμη και η Τσεχία υποδέχεται πρόσφυγες και είναι υποχρέωσή της να δείχνει αλληλεγγύη. Αλλά αλληλεγγύη πρέπει να δείξουμε και απέναντι στους συμπολίτε μας και η χρήση των ποσοστώσεων ε, δεν είναι σωστή. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει καλύτερη λύση για την εξασφάλιση των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να βοηθήσει τους πρόσφυγες ε, αντιμετωπίζοντας τα αίτια του κακού και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ασφάλειας στις χώρες προέλευσης, στις πατρίδες τους. Η κυρία Πετήρ έφυγε. Ο κύριος Κόμπερν. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε ουδής και πάνω απ' όλα εγώ μπορεί να μείνει ασυγκίνητος ε, στη θέα ενός ε, μικρού παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα. Και φυσικά ακούμε τη συνέχεια της φωνές για να δείξουμε συμπόνια. Θα πρέπει όμως να βρούμε κάποιες ε, πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα. Δεν θα με την προσπάθεια να μην σταματήσουμε, να μην αναχαιτήσουμε τη μετανάστευση που περισσότερο έχει οικονομικό χαρακτήρα, θα την αυξήσουμε και θα πολλαπλασιαστούν και οι πόλεμοι. Γιατί ε, οι χώρες του Περσικού κόλπου δεν χρηματοδοτούν τους καταβλισμούς ε, προσφύγων στην Τουρκία, στα, στα Συριακά σύνορα, για να μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στις πόλεις τους όταν δεν υπάρχει πια επίγουσα ανάγκη, γιατί τους ε, ε, ε, διοχετεύουμε προς τη Μεσόγειο για να χάσουν τη ζωή τους, αυτό είναι φρικαλαίο. Με ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών αυτών, αλλά με ενδιαφέρουν επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπατριωτών μου και το δικαίωμά τους σε μια θέση εργασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα και να πληρώσει η Μέση Ανατολή μόνη της να αναλάβει τα έξοδα αυτού του θέματος. Ο κύριος Γούλφ. Ευχαριστώ. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα έχει το δικαίωμα σε ζωή, σε τροφή, σε στέγη, σε ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση στα όρια της πατρίδας του. Κάθε άνθρωπος, ε, όταν υπάρχουν προϋποθέσεις, ε, θα πρέπει να μπορεί να μεταναστεύει σε άλλη χώρα. Βέβαια, ε, ε, οι πολίτες ε, μια συγκεκριμένη χώρα δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Και αυτές οι αρχές είναι ισχύουν για ανθρώπους σαν και εμένα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το περίπλοκο πρόβλημα της μετανάστευσης, του ασύλου και της, των προσφύγων, ελέγχοντας, προσπαθώντας να ελέγξουμε τους όρους τη μετανάστευσης Και δεν θα πρέπει μη λίγοι εκλεκτοί να, ορίζουν τις ποσοστώσεις και το, την ψαλίδα κατανομής. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στους πολίτες πόρους για να λύσουν τα προβλήματα και να μην χρησιμοποιούμε εμπριστικές, ξενοφοβικές, ρατσιστικές και εξτρεμιστικές, ε, ε, εξτρεμιστικούς χαρακτηρισμούς ε, στυλιτεύοντας κάποιους που έχουν απλώς διαφορετική γνώμη από μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα που ψηφίσαμε σήμερα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής Πόσπισιλ, αλλά δεν είναι εδώ. Μπάλτσο. Εδώ είναι, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής και συμφωνώ βεβαίω. και για το Ισραήλ και για την Παλαιστίνη υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουν όμως δεν υπάρχουν κάποια πράγματα στο ψήφισμά μας εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει να τερματιστεί η κυριαρχία του Άισις στην ε, δυτική όχθη αλλά να τερματιστεί και η συλλογική τιμωρία Πρέπει επίσης να ζητήσει την απελευθέρωση κρατουμένων και να καταδικάσει τις ε, βίες δράσεις εις βάρος επίκων. Παρά το ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός, δεν μπορώ να υπερψηφίσω αυτό το ψήφισμα. Κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει παγίως ε, την λύση των δύο κρατών. Αυτή είναι η μόνη λύση. Και βεβαίως ε, η Ιερουσαλήμ θα είναι πρωτεύουσα και των δύο κρατών και έτσι θα έχουμε ένα στιβαρό θεμέλιο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών ε, έχουν ε, ε, συναντούν συνεχώς εμπόδια. Η κυρία Μαγκερίνη πρέπει να βοηθήσει να συνεχιστούν οι συνομιλίες θα υπάρξουν ε, δύο κράτη για δύο λαούς και για όποιον άλλον θέλει να ζήσει εκεί. Κύριε Αντιπρόεδρε, όλοι άνθρωποι είμαστε και υπερτιμούμε τον κεντρικό μας ρόλο στα γεγονότα. Έτσι θεωρούμε ότι η μεταναστευτική ε, κρίση είναι δική μας ευθύνη και όχι του Άσαντ και του Ισλαμικού κράτους. Και έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να λύσουμε και την κρίση του Μεσανατολικού. Η πραγματικότητά μας είναι πως η, επιρροή, η πραγματικότητα είναι πως η επιρροή μας είναι περιορισμένη. Οι άνθρωποι εκεί της περιοχής πρέπει να επιτύχουν συμφωνία και πηγαίνουν προς τα εκεί και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και κάποιες ανταλλαγές εδαφών. Οπότε δεν έχει νόημα να έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αδέξια να λέει σύνορα του 1967. Μα αφού είναι υποδιαπραγμάτευση. Το ψήφισμα αυτό λοιπόν δεν θα προσφέρει τίποτα. Είναι για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα. Ε, δεν είμαστε εμείς το θέμα. Η κυρία Μορβάη απουσιάζει. Η κυρία Πετήρ δεν είναι πια εδώ. Οπότε Πάμε στο ψήφισμα για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ο κύριος Πόσπης απουσιάζει, ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκορωσία έχουν βελτιώσει τις σχέσεις τους πρόσφατα. Υπάρχουν δύο θετικές πτυχές στην έκθεση. Αυτό που αναφέρει για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και θετική στάση όσον αφορά την κρίση στην Ανατολική Ουκρανία βελτίωση σε σχέση με παλιές θέσεις. Είδαμε κατά τεάτια του έτους κάποιες εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφύγει μια ψύχρανση των σχέσεων. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Να συνεχιστεί η συνεργασία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα στα χέρια της Λευκορωσίας, θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε. Διότι νομίζω ότι μαζί μπορούμε να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον. Ο κύριος Χάναν, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, η Λευκορωσία αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση, όπως τη Ρωσία και την Ουκρανία με ορολογία του 1 ου αιώνα έχουμε τους Λευόφιλους και τους Δυτικόφιλους και διαφωνία. Και αυτοί που είναι υπέρ της Δύσεως δεν ανεβαίνουν σε ισχύ. Η Λευκορωσία αποφάσισε να ακολουθήσει την αυτο, ε, μια αυτοδιάθεση, αυτοκυβέρνηση και κεντρική ε, ε, κυβέρνηση και αυτονομία. Πρέπει να δεχτούμε ποια είναι τα όρια μας και τι μπορούμε να επηρεάσουμε. Πέρα του να δείχνουμε ότι υπάρχει ένα καλύτερο μοντέλο που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα για τη Λευκορωσία. Θα ήθελα να σας εξηγήσω το πώς ψήφισα για την τροπολογία 1. Στην τροπολογία αυτή εκφράζονται οι ανησυχίε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου και ζητά από τη Λευκορωσία να σταματήσει την κατασκευή μέχρι ότου ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είμαι υπέρ τη ιδέα ότι κάθε χώρα έχει αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίσει για τι ενεργειακέ πηγέ. Υπάρχουν όμω δύο σημαντικά θέματα εδώ. Καταρχήν δεν του ζητούμε να σταματήσουν την κατασκευή τελεία και παύλα, απλώ να διεξαγάγουν ανεξάρτητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γιατί η δημιουργία πυρηνικού αντιδραστήρα έχει σημαντικέ συνέπειε. Δεν είναι σαν να ε, διορθώνουμε λίγε τουρμπίνε ή ένα ηλεκτρικό εργοστάσιο. Μπορεί ένα πυρηνικό ατύχημα να ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό ζήτησα να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην επόμενη έκθεση της Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ ε, με πρώτη ομιλήτρια την κυρία Χάρκιν. Ψήφισε υπέρ της έκθεσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία. Οι μισές επιχειρήσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απασχολούν 14 εκατομμύρια ανθρώπου είναι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, που συμβάλλουν τα μάλα και στην απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στην περιβαλλοντική προστασία. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα χρήζει περισσότερη υποστήριξη. γιατί σώσαμε τις ε, ε, επιχειρήσεις τι κερδοσκοπικές, αλλά τις μη κερδοσκοπικέ δεν τις βοηθάμε. Θα πρέπει τις κοινωνικέ επιχειρήσεις να τι συμπεριλάβουμε στα εθνικά μεταρρυθμιστικά μα συστήματα. Επίσης, ε, απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τις ε, κρατικές προμήθειες και τις παραχωρήσει με κοινωνικά κριτήρια για να προωθηθεί κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία. Και επίσης, να προσυμμεθούν συγκεκριμένε ε, συμβάσει ε, για να, ε, στηριχθούν οι λιγότερο προνομιούχοι στην πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Επίσης, πρέπει να επιτρέψουμε στις κοινωνικέ επιχείρησεις να έχουν πρόσβαση στην κοινωτική χρηματοδότηση. Ο κύριος Μάμεκινς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα δυστυχώς λειτουργεί ως λειτουργεί ε, πάρα πολύ σπάνια. Δεν υπάρχει επίσης ένα σαφής ορισμός. Τι είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτό πρέπει η Κομισιόν να στηρίξει ε, τέτοιες επιχειρήσεις που εργάζονται δηλαδή κοινωνικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη στη Λετωνία. Εμείς ξέρουμε λίγα πράγματα σχετικά με αυτό. Γι' αυτό είναι λογικό νομίζω να ζητήσουμε από την Κομισιόν να επιτύξει μεγαλύτερη ε, πρωτοβουλία για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους ε, που έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μορβάη δεν είναι εδώ. Η κυρία Πετήρ ούτε αυτή είναι εδώ. Περνάμε τώρα στην τελευταία έκθεση της κυρίας Ντλαμπάγιοβα και ο κύριος Χάρκιν δεν είναι εδώ. Κύριε Χάρκιν. Η κυρία Χάρκιν, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, με χαρά το στήριξα αυτή την έκθεση. Είναι πολύ εκτεταμένη και βεβαίω αφορά το πώς θα έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας και θα ταιριάξουν ε, οι δεξιότητες με τις δουλειές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο γρήγορη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας, να μπορούμε να προβλέπουμε τις εξελίξεις ε, να δούμε τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα. Και βεβαίως να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ε, κυρίως σκεπτόμενοι πρώτα απ' όλα για αυτούς στην νομοθεσία μας. Και χάρηκα ιδιαίτερα που τα υπερψήφισε όλα αυτά το Κοινοβούλιο. Και βεβαίως είναι ένα οριζόντιο θέμα. Η έκθεση αυτή επίσης τονίζει πως πρέπει να στηρίξουμε περιθωριοποιημένες ομάδες, ανάπηρους, ε, νέους, ηλικιωμένους, ε, για να έχουν αξιοπρεπή εργασία. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκονζάλες. Εγώ ψήφισα κατά της έκθεσης, γιατί προσφέρει παλιές συνταγές που ξέρουμε ότι είναι αναποτελεσματικές και απλώς δημιουργούν ανασφάλεια, αστάθεια, φτώχεια των εργαζομένων και ανισότητα. Όταν μιλούμε για κινητικότητα, τι σημαίνει κινητικότητα, μετανάστευση. Σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν τις βαλίτσες τους και να εγκαταλείψουν για πάντα τη χώρα τους, να ξεριζωθούν. Αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η οριστική λύση για την ανεργία. Αυτή είναι η λύση για την ανεργία, η περιφέρειες που έχουν περισσότερο πληγή από την κρίση να χάνουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους που είναι τόσο δύσκολο να το δημιουργήσουν. Όταν μιλούμε για ελαστικότητα ουσιαστικά μιλούμε για εποχιακή απασχόληση, για μερική απασχόληση, για επισφαλείς θέσης απασχόλησης. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι συμπολίτε μας δεν είναι αρκετά ελαστικοί, δεν είναι αρκετά ευέλικτοι, δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και τις δεξιότητες, ότι δεν έχουν απασχολησιμότητα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς καταστρέφουμε τις θέσεις εργασίας, εμείς καταστρέφουμε τις κρατικές επενδύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε σημαντική στροφή στις οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στροφή 180 μοιρών. Ευχαριστώ. Κύριος Μάμικινς. Αγαπητοί συνάδελφοι, λαμβάνοντας υπόψη την παράδοξη κατάσταση στην Ευρώπη με τη γύρανση του πληθυσμού, μπορούμε να αναπτυχτούμε μόνο με αύξηση παραγωγικότητας Χρειαζόμαστε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, καινοτομία, κοινωνικό διάλογο, δημιουργία νέων θέσεων εργασία, θέλουμε κινητικότητα των εργαζομένων. Υποστηρίζω πλήρως τα όσα αναφέρει η έκθεση. Στηρίζω τις προτάσεις της για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε σωστές προβλέψεις. Πώς θα επηρεάσει η τεχνολογία την αγορά εργασίας. Πώς θα αλλάξει η ζήτηση όσον αφορά την αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Στο μέλλον μπορούμε να προσαρμόσουμε δεόντως όλα μας τα συστήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση να λυθούν τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Σορτζόμπο δεν είναι εδώ. Ο κ. Χάναν απεχώρησε η κυρία Μορβάη και εκείνη απεχώρησε. Άρα, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως θα προωθηθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στις αρχές της επόμενης ε, Συνόδου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα στείλω τα εγκριθέντα ψηφίσματα στους φορείς που αναφέρονται. Ολοκληρώνονται οι εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. Γεια